όχι Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε τη συνεδρία της Επιτροπής μας. Να σας ενημερώσω ότι το σημείο υπαριθμών 6 της σημερινής διάταξης αναβάλλεται Λογικά θα το έχετε λάβει και στο ενημερωτικό φυλάδιο της Κοκομπού. Ε, το... Η συνεδρίαση μεταδίδεται σε web streaming. Κάθε φορά που ανοίγετε το μικρόφωνο σας λοιπόν θα ηχογραφείτε αυτό που λέτε. Σας υπενθυμίζω ότι πρέπει να έχετε φέρει μαζί σας και τις κάρτες σας διότι θα ψηφίσουμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Να σας πω ότι η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θα κάνει ένα σεμινάριο με τα μέλη των ε, ε, Κοινοβουλίων των Δυτικών Βαλκανίων στις 23 ε, το απόγευμα και στις 24 Μαρτίου το πρωί και ο Αντιπρόεδρος Οντί θα παραστεί εκ μέρους Επιτροπής μας. Στις 23 Μαρτίου η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων μαζί με άλλες επιτροπές, μεταξύ των οποίων και η δική μας, θα κάνει μια ανταλλαγή απόψεων με τη Βαρόνη Άστον, που είναι Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα συζητήσουμε τα αποτελέσματα του, ε, του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 22ης και 23ης Μαρτίου. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, θα ήθελα να περάσω τώρα στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Τα πρακτικά τα θεωρούμε εγκριθέντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Ε, απαλλαγή 2008, 7ο, 8ο, 9ο και 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπταξης. Ο 8 9 και 10 ο ευρωπαικο ταμειο αναπταξης ο λογος στην κυρία Γιάλα Σέντερ. Παρακαλώ. Ναι, έφευρε. Όσον αφορά στο φάκελο με την ε, απαλλαγή για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης 7, ε, 8 και 9 για το 2007 Αν οι συνάδελφοι έχουν τον κατάλογο των ψηφοφοριών, θα δείτε ότι έχω διατηρήσει σε γενικές γραμμές και προσπάθησα στο μέτρο του δυνατόν να εισαγάγω και να συμπεριλάβω τις προτάσεις σας, τις προτάσεις τις οποίες θεωρούσα ότι είναι οι πλέον επικοδομητικές. Είναι αλήθεια ότι σε κάποιες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στην τροπολογία 1 της κυρίας Ανδρέασεν, ε, λυπάμαι πολύ, αλλά δεν θα μπορέσω να τη δεκτώ. Να δεκτώ δηλαδή την πρότασή σας να καθυστερήσει η απαλλαγή, διότι θεωρώ ότι οι προσπάθειες που έχει κάνει η Επιτροπή μας και που έχει αναγνωρίσει και το ελεγκτικό συνέδριο, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζουμε ότι μένει ακόμα πολλής δρόμος μπροστά μας, καταδεικνύει ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε μια αποτελεσματική διαδικασία. Κατόπιν, την πλειονότητα των τροπολογιών της κυρίας Χολμέγερ τις θεωρώ πολύ επικοδομητικές, τις έχουμε σχολιάσει και στο παρελθόν σε διάφορες συνεδριάσεις και θεωρώ ότι προσθέτουν κάποιες πτυχές, όπως για παράδειγμα την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για την Αφρική, Ε, την οποία εγώ δεν είχα συμπεριλάβει στην εκθεσή μου. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή προσθήκη λοιπόν και τα υπόλοιπα στοιχεία ε, σε γενικέ γραμμές ό,τι δεν υπήρχε το έχω λάβει υπόψη. Τώρα για τις τροπολογίες του κυρίου Σμιτ προσπάθησα να καταλάβω ποιο ήταν το σκεπτικό του και τι προσπαθούσε να μας προτείνει αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπόρεσα να τα συμπεριλάβω, διότι οι περισσότερες από τις προτάσεις τους δεν θεωρούσα ότι συνεισφέρουν στην βελτίωση του κειμένου. Ήταν μια διμερή τοποθέτηση. Καταλαβαίνω ότι η χώρα του, η, η Σουηδία έχει συγκεκριμένα προβλήματα και οι διμερείς αποφάσεις που διαθετούνται από κάποιο κράτος μέλος είναι καθόλου ένομες και αποδεκτές, αλλά σε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς εδώ, δηλαδή να πάμε λίγο παραπέρα και να εντοπίσουμε τη δυναμική της αναπτυξιακής βοήθειας από κοινοτικής πλευράς, η οποία είναι αρκετά περίπλοκη από μόνη της, είναι πολύ σημαντική και όλα όσον αφορούν στον έλεγχο των κοινοτικών δαπανών, καλό θα ήταν να τα διατηρήσουμε στην κοινοτική διάσταση και από εκεί και πέρα, ναι με ενδεχόμαστε ότι μπορεί να υπάρχουν και κάποια διμερή στοιχεία με κάποια χώρα και λαμβάνονται συγκεκριμένες αποφάσεις για τον προπολογισμό δίμερος, αλλά δεν μπορώ να δεκτώ ότι θα εισαχθούν σε αυτή τη ε, ε, διαδικασία ελέγχου του προπολογισμού και μάλιστα όταν μιλάμε για τόσο συγκεκριμένες διμερείς πτυχές. Προσπάθησα σε κάποιο βαθμό να αναγνωρίσω αυτά που έκανε ο κ. Χολμέγερ, όπως για παράδειγμα στην τροπολογία 18 ή στο εκτιμώντας 22, αλλά δεν γινόταν πλήρως. Τώρα, για την πρόταση γνωμοδότησης των ε, συναδέλφων από την Επιτροπή Ανάπτυξης. Προσπάθησα σε λογικά πλαίσια, διότι αυτό το οποίο προσπάθησαν να μας δώσουν είναι περισσότερο επί της ουσίας της ίδιας της ανάπτυξης. Προσπάθησα λοιπόν να τα συμπεριλάβω στο μέτρο του δυνατού αν υπάρχει κάποιο benchmark το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι πιο περίπλοκο να συμπεριλάβει, ε, δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Έγιναν κάποιες συζητήσεις όμως, όπως για παράδειγμα σε θέματα παιδείας, που μας επέτρεψαν να προχωρήσουμε λίγο περαιτέρω. Γι' αυτό λοιπόν προς το παρόν θα προτιμούσα να παραμείνουν οι προτάσεις των ε, ε, συναδέλφων από την Επιτροπή Ανάπτυξης, διότι θεωρώ ότι βελτιώνουν την ποιοτική πτυχή που ορισμένες φορές ε, δεν είναι τόσο προφανής σε θέματα ελέγχου του προπολογισμού. Υπάρχουν και κάποιες προφορικές τροπολογίες που θα τις δείτε στην, στον κατάλογο των ψηφοφοριών που θα ήθελα να σας ζητήσω να δεκτείτε ε, διότι προσπαθούν να βελτιώσουν κάποιες από τις πτυχές τις οποίες δεν είχαμε λάβει υπόψη. Και δέχομαι και τις τροπολογίες, ε, όπως για παράδειγμα την τροπολογία 4, δέχομαι την πρόταση της συναδέλφου της κυρίας Χολμάγερ, αλλά θα ήθελα να αναγνωρίσουμε και την ανάγκη ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να έρθει εδώ στην Επιτροπή μας το συντομότερο δυνατόν. Νομίζω ότι αυτό είναι συμπληρωματικό σε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Αυτά προς το παρόν. Ε, νομίζω ότι μέχρι τώρα ήταν πολύ επικοδομητική όλη η διαδικασία. Ο διάλογος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ε, πολύ καλός. Να τους ευχαριστήσω για την διαθεσιμότητά τους, για να μου δώσουν όλα τα στοιχεία και τη συνεργασία τους, ε, κυρίως στις πιο δύσκολες στιγμές και να ευχαριστήσω και πάρα πολύ τους συναδέλφους για τις προτάσεις τους, διότι η πρόθεσή τους ήταν να βελτιώσουν την έκθεσή μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σμίτ έχει ζητήσει το λόγο. Μπορώ να πάρω το λόγο. Ευχαριστώ την κυρία Σέντερ για την ε, έκθεσή της. Εγώ ρώτησα ένα απλό πράγμα. Γιατί απορρίψατε την τροπολογία 11, 14 και 17 και δεν μου δώσατε απάντηση. Τι λένε αυτές οι τροπολογίες. Ε, να, η Ευρωπαϊκή Ένωση να εστιάσει στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό λένε και είμαι έκπληκτος. Ε, ε, με ξαφνιάζει πώς ακριβώς, ε, για ποιο λόγο μπορεί κάποιος να απορρίψει τέτοιες τροπολογίες και δεν κατάλαβα την να έχετε επιχειρηματολογία. Είπατε όχι, δεν γίνεται, αλλά τι εννοείτε. Κοιτάξτε κύριε Σμιτ, δεν απορρίπτω το γεγονός ότι αναγνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις διάφορες χώρες και στις διάφορες περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει αναπτυξιακή βοήθεια. Και αυτό άλλωστε είναι και τμήμα της έκθεσής μου. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι περιπτώ δεν να το αναφέρουμε. Αυτό που απορρίπτω στις ε, τροπολογίες σας είναι το γεγονός ότι σε κάποιες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα όταν ε, επικαλείστε το θέμα της δημοκρατίας, δεν ξέρω τώρα, δεν τη βρίσκω την τροπολογία σας. Κάποιες από τις χώρες με τις οποίες ε, συνεργάζεται με μη κυβερνητικέ οργανώσεις και με τις οργανώσεις επιτόπου για ανθρωπιστική βοήθεια και αναπτυξιακή βοήθεια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, δεν μπορούμε να απαιτούμε το ίδιο επίπεδο δημοκρατίας το οποίο απολαμβάνουμε εμείς εδώ στην Ευρώπη. Υπάρχει μια συζήτηση για να βελτιωθεί η κατάσταση, το ίδιο και όσον αφορά στην ελευθερία έκφρασης ε, ή και σε αυτό το οποίο πολύ σωστά λέτε εσείς, ναι, μεν στην τροπολογία 11, ότι υπάρχει περίπτωση κάποιου είδου πολίτη ο οποίος βρίσκεται υποκράτηση κλπ. Αλλά και εγώ ξέρω δύο Ισπανούς που βρίσκονται σε ανάλογες ε, ή και πιο περίπλοκες συνθήκες σε άλλη χώρα, αλλά δεν είναι δυνατόν σε μια διαδικασία απαλλαγής του προπολογισμού για τις προηγούμενες ε, χρονιές να έχουμε ένα κατάλογο στον οποίο θα αναφέρουμε θύματα, αν θέλετε, μιας μάχης μεταξύ διαφόρων χωρών. Νομίζω ότι αυτό είναι θέμα της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ή της Επιτροπής Ανάπτυξης, αλλά δεν έχει σχέση με τον έλεγχο του προϋπολογισμού. Και όσον αφορά στις πτυχές ελέγχου, για την βοήθεια, για τα προγράμματα, για τη βοήθεια μέσω προϋπολογισμού, όλα αυτά είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να αξιολογήσουμε. Τη βελτίωση της διακυβέρνησης στις χώρες αυτές, ε, τη βελτίωση και την αύξηση της παιδείας και των ε, υπηρεσιών υγείας, όλα αυτά τα περιλαμβάνουμε στην έκθεση. Η τροπολογία σας ε, θεώρησα ότι ήταν περιτές, διότι ούτως ή άλλως ε, η έκθεσή μου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητούν βελτίωση των συνθηκών, αλλά τον αναφέρω στο σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, παραδείγματο χάρη ένα Σουηδό πολίτη που είναι υποκράτηση αυτή τη στιγμή, ή το να απαιτούμε συγκεκριμένες ε, προϋποθέσεις δημοκρατίας ε, και να τα θέτουμε αυτά όρο εκ των όνου κάνευ, ε, θεωρώ ότι δεν θα μπορέσουν να βοηθήσουν κανέναν, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να βοηθά χώρες οι οποίες πλήττονται από τέτοια προβλήματα και κυρίως υποφέρουν οι γυναίκες σε αυτέ τι χώρε. Κάποια χώρα μέλος, όπως για παράδειγμα η Σουηδία, διέκοψε ε, την βοήθεια που παρήχε θέματα δημοκρατίας ή πολίτες γιατί είχε θέματα δημοκρατίας ή ε, πολίτες σε κάποια δύσκολη κατάσταση, πολίτες υποκράτηση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλα αυτά θα διέπουν την κοινοτική πολιτική. Ε, η οποία κοινοτική πολιτική έπρεπε, έρχεται ως συμπλήρωμα ή ως ε, ένδειξη, αν θέλετε, των συμπληρωματικών διμερών ε, πολιτικών. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να αναφερόμαστε σε τέτοιες συγκεκριμένες παρεπτώσεις οι οποίες αναφέρονται στις διμερείς σχέσεις που έχει αυτή τη στιγμή η Σουηδία για τη βοήθεια που παρέχει ως Σουηδία σε συγκεκριμένες χώρες. Ευχαριστώ. Πρέπει να, ψηφίσω, κύριε ε, να ψηφίσουμε κύριε Σμιτ γρήγορα. Ε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, Πρόεδρε. Για την 11 συμφωνώ, αλλά για τις 14 και 17 διαφωνώ. γιατί νομίζω κάνετε λάθος με τα επιχείρηματα που προβάλλετε. Money talk λέμε στα αγγλικά, ότι αυτό που ε, είναι το σημαντικό για όλους είναι τα χρήματα ε, και νομίζω ότι αυτό ισχύει και σε συγκεκριμένη περίπτωση. Ωραία. Να περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία. Έχετε όλη την κάρτα σας για να ψηφίσουμε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Ψηφίζουμε την πρόταση απόφαση για την απολαγή. Έχουμε την τροπολογία 1 που παρουσίασε η κυρία Ανδρέασαν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 18 ψήφοι κατά 3 υπέρ. Περνάμε τώρα στην απόφαση για απαλλαγή στο σύνολό της, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας. 19 voti 2 contrari. Εγκρίνεται 19 υπέρ, 2 κατά. Να περάσουμε τώρα στην πρόταση απόφασης για το κλείσιμο των λογαριασμών στο σύνολό τους. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 19 ψήφοι υπέρ, 3 κατά. Να περάσουμε τώρα στην προφορική τροπολογία υπαριθμών 1. Άρχεται η ψηφοφορία. La votazione... Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 19 ψήφοι κατά, 3 υπέρ. Ψηφίζουμε την τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 21 ψήφοι υπέρ, μία αποχή. Τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 12 ψήφοι υπέρ, 10 κατά. Περνάμε τώρα στην τροπολογία Προφορική τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 17 ψήφοι υπέρ, 3 κατά, μία αποχή. Τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 16 ψήφοι κατά, 5 υπέρ, μία αποχή. Τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 19 ψήφοι κατά, 3 υπέρ. Τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας εγκρίνεται 14 ψήφοι υπέρ, 8 κατά. Τροπολογία 8. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 19 ψήφοι κατά, 3 υπέρ. Τροπολογία 1 της Επιτροπής Ανάπτυξης. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 22 ψήφοι υπέρ. Τροπολογία 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 19 ψήφοι υπέρ, 3 κατά. Τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη εγκρίνεται. 22 ψήφοι υπέρ. Τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 17 ψήφοι κατά 4 υπέρ. Τροπολογία 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 23 ψήφοι υπέρ. Τροπολογία 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. 13 ψήφοι υπέρ, 9 κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 14, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 14 ψήφοι υπέρ, 8 κατά. Τροπολογία 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίνεται 12 ψήφοι υπέρ, 9 κατά. Τροπολογία 6 της Επιτροπής Ανάπτυξης. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορίας. εγκρίνεται 23 ψήφοι υπέρ. Προφορική τροπολογία υπαριθμών 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 23 ψήφοι υπέρ. Τροπολογία 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 17 ψήφους κατά, 5 υπέρ και μία αποχή. Τροπολογία 18. Ε, άρχεται η ψηφοφορία, συγγνώμη. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 23 ψήφους. Τροπολογία 3. Ε, επιτροπή Ανάπτυξης. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 23 ψήφους. Τροπολογία 7 της Επιτροπής Ανάπτυξης. Άρχεται η ψηφοφορία, πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 23 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 4 τη Επιτροπής ανάπτυξη. άρχεται η ψηφοφορία, πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 23 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας εγκρίνεται με 21 ψήφους υπέρ, 2 κατά. Προφορική τροπολογία 4, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 23 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 21, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 23 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 22, άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 23 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 23, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασης ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 23 ψήφους υπέρ τροπο, προφορική τροπολογία υπαριθμών 5, άρχεται η ψηφοφορία, Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 21 ψηφί υπέρ. Έχουμε τώρα την τελική ψηφοφορία. Ως τροποποιήθηκε το κείμενο, άρχεται η ψηφοφορία, πέρασε της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 21 ψήφοι υπέρ, 2 κατά. Ευχαριστούμε την κυρία Γιάλα Σέντερ για την δουλειά που έκανε. Και τώρα βρισκόμαστε στο σημείο 5 της μερίσιας διάταξης, ειδική έκθεση 17 του 2009 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης γυναικών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Να δώσουμε το λόγο και να χαιρετήσουμε και τον εκπρόσωπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Βίντιου Ίσπυρ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Είναι εδώ ο κύριος Οβίντιου. Thank you, Mr. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε την ευκαιρία να είμαι εδώ σήμερα το απόγευμα για να είμαι παρόν στην εξέταση αυτή ανταλλαγής απόψεων στο έγγραφο εργασίας που αφορά την ε, υπαριθμό 17 έκθεση, ειδική έκθεση του Ελεκτρικού Συνεδρίου του 2009 για την επαγγελματική κατάρτιση δράσεων γυναικών που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αυτή είναι η πρώτη ειδική έκθεση του συνεδρίου που αφορά ιδιαίτερα το θέμα της ισότητας των ευκαιριών από τότε που αποφάσισε το Κοινοβούλιο του 2007 να είναι ένα κέριο θέμα η ισότητα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Βαμ, για την σαφή και πλήρη αντιμετώπιση της έκθεσης του συνεδρίου στο έγγραφο εργασία και για την ομιλία του που ακούσαμε μόλις για το σημαντικό θέμα της επαγγελματικής κατάρτισης που η Ευρωπαϊκή Ένωση με 2006 ενίσχυσε με 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η έκθεση του συνεδρίου εξετάζει κατά πόσον έχει γίνει η σωστή επιλογή των δράσεων επαγγελματική κατάρτισης για τις γυναίκες σύμφωνα με τα κριτήρια ανάλυσης αγοράς και κατά πόσον οι πληροφορίες εποπτείας ήταν σύμφωνες με τους στόχους των ε, εν λόγω Θα ήθελα να επαναλάβω τα αποτελέσματα και συστάσεις από την, ε, τον έλεγχο για την ανείχνευση και την επιλογή των δράσεων επαγγελματική κατάσταση για τι γυναίκε, τα συμπεράσματα είναι ότι αυτέ οι δράσει στα προγράμματα που εξέτασε το συνέδριο δεν ήταν σύμφωνα με τις αναλύσεις αγοράς και με τα μέτρα που είχαν καθοριστεί και έτσι δεν εστιάστηκαν ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες ομάδες στόχους. Επιπλέον, ο τρόπος με τον οποίο τα σχέδια αυτά επελέξαν δεν ήταν σύμφωνα με τις ανάγκες της ε, αγοράς απασχόλησης και δεν εξασφάλιζαν ότι κάθε συγκεκριμένο σχέδιο θα ήταν ευθυγρασμένο με τους γενικούς στόχους των προγραμμάτων. Το συνέδριο σύμφωνα θεωρεί ότι μια ανάλυση τέτοια της αγοράς θα πρέπει να τονίζει τον καθορισμό λειτουργικών προγραμμάτων και ότι ο τύπος εκπαίδευσης που αποφασίστηκε θα πρέπει να βασίζεται πάνω στην ανάλυση αυτή. Όσον αφορά το θέμα του κατά πόσον υπήρχε καλή αξιολόγηση των επιτεύξεων και των στόχων, το ε, συνέδριο θεωρεί ότι οι πληροφορίες εποπτείας δεν επιτρέπουν μια τέτοια αξιολόγηση. Τα προβλήματα συμπεριλαμβάνουν τους δείκτες, την έλλειψη στόχευσης και την ε, υποβολή ανεπαρκών ή μη βάσιμων πληροφοριών. Κατά την άποψη του συνεδρίου, η κατάσταση αυτή δεν οδήγησε τις υπεύθυνες ε, αρχές των κρατών μελών ή και την Κομισιόν να μπορεί να κρίνει κατά πόσον οι στόχοι επιτέχθησαν ή όχι. Γι' αυτό το συνέδριο θεωρεί ότι θα πρέπει η Κομισιόν να έχει δική της μονάδα επιτήρησης, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τους σωστούς δείχτες που θα πρέπει να καθοριστούν από τα κράτη-μέλη <clears throat> για να υπάρχει η πλήρης και ε, σεβαστή ενημέρωση. Ως μέρος του ελεκτικού συνεδρίου υπεύθυνο για την έκθεση αυτή, θέλω να πω ότι ήταν πάρα πολύ καλό που ο κύριος Βόχαμ θετικά υποδέχθηκε την έκθεση και ότι σημειώσει τις αναμίες που υπάρχουν. Θεωρούμε ότι το συνέδριο θα πρέπει να λάβει υπόψη τα ευρύτερα θέματα των γυναικών που επιστρέφουν στον χώρο εργασίας και την ανάγκη βελτίωσης των ε, προσώνων τους κατανοούμε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες της αγοράς απασχόλησης, πράγμα για το οποίο προϋποτίθεται η σχετική κατάρτιση. Θεωρούμε όμως ότι θα πρέπει να περιμένουν περισσότερες δράσεις να είναι εστιασμένες, ούτως ώστε να μπορεί να οδηγήσουν στην απασχόληση. Εν κατακλείδη, θα ήθελα να σας πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος που μπορώ να είμαι σήμερα εδώ και να συζητήσω την έκθεση αυτή που έγινε θετικά δεκτή από το Κοινοβούλιο. Γενικά η έκθεση έγινε πολύ θετικά δεκτή. Πρόκειται για ένα τομέα πάρα πολύ σημαντικό για τον Ευρωπαίο πολίτη και όχι μόνο για τις γυναίκες στην κοινωνία μας, αλλά για όλους εμάς. Και γι' αυτό ελπίζω ότι η έκθεση και τα συμπεράσματα, όπως θα τα κρίνετε και ενισχύσετε κι εσείς, θα μπορέσει να συμβάλλει προς μια Ευρώπη στην οποία προσπάθειες καταβάλλονται για την προώθηση των ίσων ευχαιρών ανδρών και γυναικών στην αγορά απασχόλησης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Βόγκαν, εισηγητή. Oh, um, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο στην ιδιαίτερα που προετοίμασε την έκθεση αυτή και τον κύριο για τη συμβολή του. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική έκθεση γιατί αξιολογεί τα σχέδια τα οποία ε, χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Και ξέρουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μεταξύ άλλων στόχων προσπαθεί να καταρτιστούν εκείνοι που προσπαθούν να επανέλθουν στην αργοδά 4 δισεκατομμύρια ε, ευρώ για την περίοδο 2000-2006 ε, για τις γυναίκες. Για να μπορέσουν να προωθούν έτσι οι ισότητες των ευκαιριών. Θα ήθελα να τονίσω στους αδέλφου ότι η έκθεση αυτή θα πρέπει να εξεταστεί από κοιμού με άλλα σχέδια τα οποία χρηματοδοτούνται από τα κράτη-μέλη, γιατί βέβαια και τα κράτη-μέλη μπορούν, άμα θέλουν, να χρηματοδοτήσουν τα δικά τους προγράμματα και να παίξουν σημαντικό ρόλο εδώ. Το ελεκτικό συνέδριο θα έχει λάβει φαντάζομαι υπόψη τα κριτήρια επιλογή για τα σχέδια και για τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τα κράτη και το Κοινωνικό Ταμείο και είναι λυπηρό, όπως είπανε, ότι δεν υπήρχε αρκετή διάκριση από τα προγράμματα για γυναίκες μόνο και από άντρες και γυναίκες. Επίσης, οι πληροφορίες ήταν στη μόνο για 42% ε, των προγραμμάτων. Ή σε άλλες περιπτώσεις θεωρήθηκε ότι μία μονάδα μόνο κατάρτιση ήταν επαρκή για να θεωρηθεί ότι έχουν αποκτήσει την πλήρη κατάρτιση. Οι άλλοι δεν χρειάστηκε να αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ε, εργαστούν με πλήρη απασχόληση μετά που θα δηλώσουν την κατάρτισή τους. Αυτό είναι το θέμα της ε, ανάλυσης ε, των στόχων. Η ανάλυση του ηλεκτρικού συνεδρίου. Είναι απόλυτα λογική. Θα ήθελα όμως λιγάκι να τη σχολιάσω. παραδείγματο χάρη, θα ήθελα να τονίσω ότι αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στην ανάλυση της νέας αγοράς ε, ε, απασχόλησης και του ρόλου των γυναικών στην αγορά αυτή, παραδείγματος χάρη, όσον αφορά τις ανάγκες για ευέλικτα ωράρια, για, την, ε, για, για να μπορούν να κρατούν τα παιδιά τους κάπου Δηλαδή δεν είναι πάντα ευθυγραπονέμες οι προτεραιότητες της αγοράς απασχόλησης με τους στόχους. Ελπίζω ότι το ελεκτρό συνημερίσια τη απόψη αυτός τονίζουν επίσης ότι δεν υπάρχει αρκετή διαφοροποίηση μεταξύ των προγραμμάτων που είχαν σαν στόχο μόνο τις γυναίκες και εκείνους που είχαν άντρες και γυναίκες σαν στόχο. Θα μπορούσαμε βέβαια να πούμε ότι γενικά ο στόχος είναι και οι άντρε και οι γυναίκε να κατευθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιώσουν τι ικανότητέ του να μπορούν να συμμετέχουν στην αγορά απασχόληση. Αυτά είναι νομίζω ε, συμπληρωματικά μέτρα μέσα στα πλαίσια της, ε, του λεγόμενου mainstreaming, της εσωνάς δηλαδή τη του σε όλε τι δραστηριότητε αυτέ. Θα μπορούσα να συμφωνήσω με το ηλεκτρικό συνέδριο στο ότι χρειάζεται να βελτιωθεί η κατάσταση για να βελτιωθεί η παρακολούθηση και να υπάρχουν ξεκάθαρα στάνταρ, τονίζοντας ιδιαίτερα τον στόχο της μείωσης του χάσματος μεταξύ των δύο φύλων. Τελικά θα ήθελα να πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι ένα μέσο σε πολλές χώρες για να μπορέσουν οι γυναίκε να επανέλθουν στην αγορά εργασία με τη βελτίωση τη κατάρτισή σα. Και ελπίζω ότι το κοινωνικό τμήμα θα συνεχίσει προ την ίδια άγουσα και στο μέλλον. Θα ήθελα επίση να συμφωνήσω ότι είναι σημαντικό τα προγράμματα αυτά να βασίζονται σε μια ανάλυση αγοράς απασχόλησης, αλλά θα πρέπει να εξεταστούν και άλλα στοιχεία σχετικά. Και τέλο, θα πρέπει βέβαια να υπάρχουν οι κατάλληλοι δείκτες για τα προγράμματα, όπως είπε και το ηλεκτρικό συνέδριο. Χρειάζεται να υπάρχει καλή και αποτελεσματική επιτήρηση και εποπτεία. Με αυτά τα σχολεία θα ήθελα να πω ότι χαιρετίζω την έκθεση αυτή και να ευχαριστώ το συλλεκτικό συνέδριο για την εργασία του. ευχαριστώ κύριε Γκρέσλε. Ευχαριστώ πολύ. Μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση. Όχι μόνο επειδή επενδύουμε πάρα πολλά χρήματα, σε ειδικά προβλήματα ενίσχυση των γυναικών, αλλά και οι γυναίκε σχετίζονται και πάρα πολύ με τη στρατηγική Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής και με το θέμα το πώ θα αυξήσουμε το ποσοστό των γυναικών στην αγορά εργασία. και γι' αυτό το θέμα γυναίκα είναι πάρα πολύ σημαντικό στο πρόγραμμα και γι' αυτό απορώ πώς μπορεί σε ένα πρόγραμμα που στο στοχεύει στις γυναίκες υπάρχει ένα ποσοστό συμμετοχής ανδρών 27% όπως είναι στο πρόγραμμα αυτό στην Ιταλία. Είναι πάρα πολύ φιλόδοξο το πρόγραμμα και δεν μπορώ από τη συζήτηση να καταλάβω γιατί είναι σημαντικό να προωθηθούν οι γυναίκες στην αγορά απασχόλησης και γιατί είναι σημαντική συμβολή του κοινωνικού ταμείου. Αυτό δεν είναι σωστό όμως. Και γι' αυτό θα ήθελα να ξέρω τι θα κάνει η Κομισιόν για να βελτιώσει το αποτέλεσμα. Εγώ ασχολήθηκα συγκεκριμένα με τα μέτρα του ε, Κοινωνικού Ταμείου στη δική μου εκλογική ε, περιφέρεια. Γιατί εγώ έχω πάρα πολλές ε, γυναίκες πάνω από τα 50 μετανάστριες και θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται για να μπορώ αυτή η ομάδα του πληθυσμού να βοηθηθεί για να μπορέσει να ενταχθεί στην αγορά εργασίας. Από αυτά που άκουσα μέχρι στιγμής δεν βοηθούμε ιδιαίτερα γιατί έχουμε να κάνουμε και με το θέμα της υποδομής για τα παιδιά και όλα αυτά. Τι ξέρουμε σχετικά. Πόσο καλές είναι οι υποδομές στα κράτη-μέλη για να μπορέσει να δοθεί η δυνατότητα στις γυναίκες να εργαστούν. Ποια είναι μέχρι στιγμής η δυνατότητα συντονισμού των διαφόρων προγραμμάτων μεταξύ τους για να μπορέσει ένα κράτος μέλος να κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή. Γι' αυτό θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο το ελεκτικό συνέδριο έχει εξτάσει το θέμα αυτό. Ποιοι είναι οι όροι που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην αγορά απασχόλησης. Και κατά πόσο πραγματικά είναι χρήσιμο σε ένα κράτο μέρο να υπάρχουν αυτού του τύπου τα προγράμματα. Και θα ήθελα να συστήσω κατεπηγόντως να είμαστε πιο φιλόδοξοι, γιατί αυτό είναι ένα πρόβλημα κλειδί και για την αγορά εργασίας, αλλά και για όλους εκείνους που προσπαθούν πραγματικά να μπουν στην αγορά αυτή απασχόλησης. Ε, αυτό που με, που με ενόχλησε είναι η μικρή αηφορία των προγραμμάτων. Εγώ έχω μία εκλογική περιφέρεια με ανεργία της τάξης του 5%. εξέτασα να δω ποιες είναι οι καλύτερες πρακτικές που εφαρμόνται και βλέπω ότι ε, ε, επαρχίες ή κομμόπολεις που βρίσκονται η μία δίπλα στην άλλη δεν ξέρει η μία τι κάνει η άλλη. Και όλοι αυτοί οι μετανάστες που ίσως ε, προέρχονται από τη Ρωσία όπως εμείς εμάς κυρίως δεν ξερει η μια τι κανει η αλλη και ολοι αυτοι οι μεταναστες που ισως προκειται απο τη ρωσια οπως εμεις εμας κυριως δεν έχουν τίποτα το πιο σφαιρικό, το πιο συντονισμένο για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει, είναι, θα μπο, πρέπει να μπορούν όλοι να μάθουν μένα από τους δέα εφόσον έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις στην περιοχή. Ευχαριστώ. Θέλει να παρέμβει ο πρόσωπος του ελεγκτικού συνεδρίου. Mulțumesc pentru intervenția doamnei deputat Gresel. Θα ε, ε, ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γκρέσλε για την παρέμβασή της. Ως προς τις ερωτήσεις, νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να απευθύνει τόσο πολύ στο ελεγκτικό συνέδριο, μάλλον θα έπρεπε να τις απευθύνει στην Επιτροπή. Εμείς κάνουμε έναν έλεγχο για μία πολιετή περίοδο. Κατόπιν αίτησης του Κοινοβουλίου, λοιπόν, συντάξαμε αυτό το σχέδιο απαλλαγής και υποβάλαμε συστάσεις. Τα πορίσματα κρίνω είναι ε, σαφή. Η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών νομίζω θα συμφωνήσει με το ότι είναι σαφή τα συμπεράσματα και με αυτά τα δεδομένα μπορούμε να απαντήσουμε στην κυρία Γκρέσλε η ευθύνη μας περιορίζεται ε, στο αντικείμενο της αναλύσεώς μας. και μπορούμε να δώσουμε μια συνέχεια στο μέλλον. Είναι περίπλοκη η κατάσταση, έχει δίκιο η κυρία Γκρέσλε και δεν ε, συζητούμε εδώ μόνο για τα ταμεία ή μόνο για τα προγράμματα. Συζητούμε για τις ε, αρχές ε, που, οφείλουμε, που πρέπει να τηρούνται. για να βρεθεί απάντηση θα έλεγα ότι ακούσαμε την άποψη του ελεγκτικού συνεδρίου και τώρα είναι η σειρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δώσει κάποιες ε, απαντήσεις, να μας εξηγήσει τι θα κάνει στο μέλλον για να βελτιώσει την κατάσταση. Υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα ήθελε να παρέμβει για το σημείο αυτό. Παρακαλώ. Είμαι ο Γενικός ο διευθυντής ε, της ε, ε, μονάδας επιφορτισμένης με τον έλεγχο για τα προγράμματα ισότητας των δύο φύλων και ε, Ω προ τι διαπιστώσει του ελεγκτικού συνεδρίου δεν έχουμε καμία διαφωνία. Παρόλα αυτά θεωρούμε ότι η έκθεση αυτή εστιάζεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο. Η ισότητα των ευκαιριών είναι ε, εγκάρσιο στόχο ε, του ΕΤΑ. 78 δις περίπου για την περίοδο 2000 με 2006 και άρα είναι ε, λιγότερο από το 5% του κονδυλίου του Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο καλύπτει και μια σειρά εθνικών μέτρων για την ισότητα των ευκαιριών στην αγορά εργασία. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο με μια τόσο συγκεκριμένη έκθεση να καταλήξουμε σε ε, γενικότερα συμπεράσματα για την πολιτική, για την πρόθεση της ισότητας ε, των δύο φύλων. Σημειώνουμε τα συμπεράσματα του ελεγκτικού συνεδρίου και εν μέρη τα έχουμε λάβει υπόψη κατά την τωρινή περίοδο προγραμματισμού 2007 έως 2013 για τους δείκτες επιδόσεων παραδείγματος χάρη και τους στόχους ως προς τις ε, επιδόσεις για τα επιμέρους ε, σημεία που ανέφερε τώρα η κυρία Γκρέσλι υπάρχουν κάποια μέτρα και έχουμε πλήρη επίγνωση τη ε, βαρύτητά του για την απασχολησιμότητα των γυναικών, όπω η φροντίδα των παιδιών, παραδείγματο χάρη. Αλλά έχουμε ε, περιορισμένο περιθώριο ελιγμών στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Τι μπορεί να κάνει να συμβάλλει στις δαπάνες ε, για τους ε, βρεφονιπιακούς σταθμούς όταν παρακολουθούν κάποια κατάρτιση οι γυναίκες παραδείγματος χάρη αλλά κατά τα λοιπά δεν μπορεί να παρέμβει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και παρότι αναγνωρίζουμε τη βαρύτητα αυτού του σημείου. Για τους άντρες τώρα όπως διαπίστωσε και το ελεγκτικό συνέδριο Πρέπει να ερμηνεύσουμε με κάποια ευελιξία τους κανόνες γιατί προσάπτουμε υπερβολική αυστηρότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορισμένε φορές. Ε, λοιπόν υπήρχαν δράσεις κατάρτισης ε, που είχαν προετοιμαστεί με ένα συγκεκριμένο αριθμό θέσεων αλλά ε, δεν καλύφθηκαν όλες οι θέσεις. Οπότε οι διοργανωτές δέχτηκαν και κάποιους άντρες. Νομίζω ότι είναι σωστή η διαχείριση γιατί πρέπει στο έπαιρμα να αξιοποιούμε τα διαθέσιμα μέσα. Δηλαδή να αφήνουμε ανεπρόσδεκτες θέσεις μόνο και μόνο επειδή δεν υπήρχαν αρκετές γυναίκες. Για το μέλλον τώρα, πολλέ συστάσει του ελεγκτικού συνεδρίου ήδη έχουν ε, συμπεριληφθεί στην τωρινή περίοδο προγραμματισμού και η Επιτροπή έχει δρομολογήσει τη συνολική αξιολόγηση τη προηγούμενη ε, περίοδου, το 2006, ε, και θα κοινοποιηθεί το αποτέλεσμα φυσικά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από αυτή τη βάση θα προετοιμάσουμε τα νέα μέτρα για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού και θα έχουμε και τα αποτελέσματα του χρόνου κατά πάσα πιθανότητα. Ευχαριστούμε κυρία Σάντε. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ για να κατανοήσω λίγο καλύτερα το σύστημα αξιολόγησης αυτών των προγραμμάτων και εδώ να πω ότι συμφωνώ απολύτως ε, με την κυρία Γκρέσλερ ότι είναι θεμελιώδη σημασία, μα ενδιαφέρουν πολύ και πράγματι θα μπορούσαν να βοηθήσουν τι γυναίκε να τοποθούν, καλύτερα στου τομεί στου οποίου δεν είναι παρούσε. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τον κύριο Βόγκαν. Στο κείμενο που έχουμε εδώ, δεν έχω ακόμα δει το CD, οπότε μιλάω για το κείμενο, για το έγγραφο μας έχετε δώσει. Στην ε, σελίδα 5 σχολιάζεται δύο προγράμματα τα οποία εμφανίζονται μετά από την αξιολόγηση. Και λέτε ότι για την περίπτωση του προγράμματος Λομπάρντο διαπιστώνεται ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, διότι για τις νέες γυναίκες ε, για τις οποίες υπήρχε πρόθεση κατάρτισης, υπήρχε πρόβλημα στις, στην αγορά εργασίας. Θα ήθελα να ξέρω αν αυτό είναι δική σας άποψη ή απροκύπτει από τις γυναίκες οι οποίες ε, ε, απέκτησαν θέση εργασίας αμέσως. Το να είναι κάποιο, για παράδειγμα, μία νέα γυναίκα άνεργη σε χώρες όπως τη ε, δική μου, για παράδειγμα, ή την Ιταλία, δεν σημαίνει ότι έχει μία πάγια θέση στην αγορά. Ίσα ίσα πολλές φορές πρέπει να ανακυκλώσουμε αυτές τις νέες, γιατί πρόκειται κυρίως για νέες γυναίκες και να τους προσφέρουμε περισσότερες εγγυήσεις ότι θα βρουν μια θέση εργασίας, ακόμα και αν δεν είναι ανάλογο των δυνατοτήτων τους, αλλά τουλάχιστον να είναι μια θέση εργασίας. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν αν αυτή η δήλωση είναι δική σας, προέκυψε από την αξιολόγηση ή προκύπτει από το πρόγραμμα. Επίσης, για το πρόγραμμα για την Ανταλουσία, όπου λέτε ότι τα προγράμματα αυτά, τα ε, χρήματα τα οποία διατίθενται δεν ε, ε, βολεύουν, αν θέλετε, τις γυναίκες που ασχολούνται και με τα παιδιά τους. Ε, δυστυχώς στην Ανταλουσία έτσι έχει κατάσταση. Οι περισσότερες γυναίκες ε, δεν είναι σε θέση να ε, στήριζονται στον σύζυγό τους, πρέπει οι ίδιες να φροντίζουν τα παιδιά τους. Επομένως, ε, θα ήθελα να ξέρω το ωράριο εργασίας που αναφέρεται εδώ είναι κάτι το οποίο προέκυψε με λόγο αξιολόγησης, το ακούστε από τις ίδιες τις γυναίκες ή είναι δική σας άποψη. Και τέλος, λέτε ότι υπάρχουν κάποια προγράμματα στα οποία έχουμε καθορίσει πολύ καλά ποιες γυναίκες θα συμμετέχουν, αλλά εδώ έχει και κάτι το οποίο δεν συνάδει με τα υπόλοιπα ήταν άνεργες 3 με 12 μήνες μετά την κατάρτιση. Μετά από την προηγούμενη κατάρτιση που έχουν λάβει ή από την κατάρτιση από το Κοινωνικό Ταμείο. Αυτά θέλω να μου τα διευκρινίσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βόγκαν θέλει να απαντήσει στις ερωτήσεις της κυρίας Σέντερ. Yes, uh, ναι, ναι, πρόεδρε, ευχαριστώ. Τα θέματα που έδειξε η κυρία Σέντερ είναι θέματα διαδικαστικά και ίσως το ηλεκτρικό συνέδριο να απαντήσει καλύτερα. Αλλά θα αναφερθώ σε κάποια δύο-τρία θέματα. Δυστυχώς η κυρία Γκρέσλα έφυγε και αναφέρθηκε στο θέμα της συμμετοχής 20% ανδρών σε κάποια από τα προγράμματα αυτά. Αυτό βέβαια το είδαμε πραγματικά σαν ένα σημαντικό θέμα, το εξέτασε και το ηλεκτρικό συνέδριο έτσι. Τώρα δεν ξέρουμε κατά πόσον ποια είναι η καλύτερη λύση είναι απλώς mainstreaming, μεγαλύτερη συμμετοχή δηλαδή, ή εστιασμένη και ειδικά αποκλειστικά μόνο γυναίκες. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι λόγω δείκτες εδώ υπάρχουν και ότι το θέμα της παρακολούθησης και εποπτείας είναι επίσης σημαντικό γιατί έτσι μονάχα μπορούμε να αξιολογήσουμε την επιτυχία των σχεδίων και αυτό είναι έτσι ένα σημαντικό έργο της Κομισιόν και θα πρέπει να το λάβει υπόψη μετά τη δημοσίευση αυτής της έκθεσης. Και χάρηκα που η κυρία Γκρέσλε συμφωνεί μαζί μου για τη σημασία άλλων θεμάτων. Θα το θίξω αυτό στην έκθεσή μου. Η ανάλυση δηλαδή της αγοράς εργασίας δεν συμπίπτει πάντα με το τι είναι καλύτερο για τις γυναίκες. Αυτά τα θέματα πρέπει να τα εξετάσουν και άλλοι συνάδελφοι όπως και εγώ έθιξαν αυτό το θέμα και ελπίζουμε γι' αυτό ότι στο ηλεκτρικό συνέδριο οι υπεύθυνοι για το σχέδιο αυτό θα το έχουν κατά νου για το μέλλον. Και τέλος θα ήθελα να σας πω ότι η χρηματοδότηση του Κοινωνικού Ταμείου σε πολλά μέρη ήταν πάρα πολύ θεματική και γι' αυτό θα πρέπει εξτάσω στην έκθεση αυτή και κοιτάζω τι θα κάνουμε στο μέλλον να είμαστε σίγουροι ότι η χρηματοδότηση είναι επιτυχής. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ τον κύριο Βόγκαν. Τώρα, επειδή ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση, θα ήθελα να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά λάβαμε μία επιστολή η οποία είχε αποστολέ εμένα από τον Υπουργό Εξωτερικών Επιθέσεων της Ουγγαρίας για το θέμα του διορισμού του μέλους του ελεγκτικού συνεδρίου του κυρίου Φάτσακας φρόντισαν να δοθεί αντίγραφο αυτής της επιστολής σε όλους τους ε, ε, συντονιστές. Λύεται η συνεδρίαση μέχρι αύριο στις 9 το πρωί. Αύριο το πρωί έχουμε μία πληρέστατη ημερήσια διάταξη. Καλησπέρα σε όλους.